E λοιπόν, συνάδελφοι, συνεχίζουμε τις ψηφοφορίες. Έκθεση Μάριο Ντάβιτ και Μάρεκ Σίβιετς για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας. Δεν έχουμε τροπολογίες, ψηφίζουμε ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές, δεκτή. Συγχαρητήρια στους δύο εισηγητές. Έκθεση της κυρίας Ίντβελντ σχετικά με την αντιτρομοκρατική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ψηφίζουμε την πρώτη τροπολογία. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ε, ψηφίσουμε ηλεκτρονικός. Άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν ε, άπαντες. Έληξε ψηφοφορία. Έγινε δεκτή η ε, τροπολογία πρόταση ψηφίσματος καταπίπτει ως εκ τούτου ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίε Καλή σα όρεξη και θα περάσουμε στις επεξηγήσεις ψήφου.